So uh, Καλησπέρα σας κύριοι συνάδελφοι. Σας καλωσορίζω στην, στο δεύτερο μέρος. Ελπίζω να φάγατε καλά και δροσιστικά. Το απόγευμα θα μιλήσουμε για το θέμα των εσωτερικών-εξωτερικών, κυρίως όμως των εξωτερικών, στον τομέα της ελευθερίας, δικαιοσύνης κλπ. Σας θυμίζω ότι το πρωί πολύ στα παραδείγματα που αναφέρατε, είπατε με τι ανθρω... προβλήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων ασχολείστε στις χώρες σας όπως τους μετανάστες. Είναι θέματα που και εμείς τα συζητούμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Επιτροπή Εσωτερικών ακριβώς. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε προβλήματα και προκλήσεις και σε ολόκληρη την Ένωση μέσα, στο εσωτερικό της και σε κάθε χώρα. Όταν γίνονται πολυμερείς συνεννοήσεις ή συζητούμε με συναδέλφους από χώρες εκτός της Ένωσης, δεν θα είμαστε αξιόπιστοι αν δεν ασχοληθούμε και με τα του οίκου μας. Γι' αυτό λοιπόν θέλουμε να ακούσουμε και από εθνικής πλευράς, από εσά δηλαδή, με ποιο τρόπο θα μπορούσαμε να τα λύσουμε όλα αυτά συνεπέστερα. Πριν δώσω το λόγο στον πρόεδρο της Επιτροπής Δημοσίων Ελευθεριών θα ήθελα να σας καλέσω αν μπορείτε να μείνετε παραπάνω γιατί μετά τη συνεδρίαση στο, στην ίδια αίθουσα σήμερα οργανώνεται ακρόαση για την πολιτική των επανεισδοχών και τις επιπτώσεις της επί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μπορεί να σας ενδιαφέρει μερικούς. Και τώρα Χαίρομαι για την παρουσία του κυρίου Χουάν Φερνάντε Λόπε Αγγιλάρ που είναι πρόεδρος τη Επιτροπής Δημοσίων Ελευθεριών, δικαιοσύνη και Εσωτερικών. Γιατί έτσι θα δει, φαίνεται ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα τα συνδυάζουμε και με τα εξωτερικά θέματα και με τα εσωτερικά. Πριν όμως του δώσω το λόγο, θα ήθελα να σας παρουσιάσω τους εμπειρογνώμενους Μόρσομ Κύρων που είναι διευθυντής του Ιδρύματος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Ένωσης από τη Βιέννη και η κυρία Φιγκάντε Μιλασιούτε που είναι πρόεδρος του Τμήματος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και λοιπά του Συμβολίου. Ορίστε κύριε Αγγιλάρ μου. Σας ευχαριστώ κυρία Τσέρ, κυρία Μπαρβάρα Λόχμπιλε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς που είναι παρόντες. Είμαι εξόχως ευτυχισμένος που μπορώ και πάλι να είμαι παρόν σε αυτή την εκδήλωση συνεργασίας μεταξύ Κοινοβουλευτικών Εθνικών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και μεταξύ Επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Επιτροπής της οποίας προείσταμε, Επιτροπής Δημοσίων ελευθεριών και θεμελιωδών δικαιωμάτων. Έχουμε συζητήσει πολύ συχνά αυτά τα θέματα του σχεδίου δράσης Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα που είναι και το κεντρικό θέμα της σημερινής συζήτησης. Ο στόχος μας πρέπει να είναι να εξασφαλίσουμε την εσωτερική και εξωτερική συνεκτικότητα της ευρωπαϊκής πολιτικής για τα ανθρώπινα δικαιώματα και η συνεργασία από την πλευρά των, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου των Επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απαιτεί σημαντική προσπάθεια. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης την εφαρμογή των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων με έναν τρόπο που διαπνέεται από την δέσμευσή μας στα οικουμενικά ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δίκαιου, το αδιέρετο των θεμελιωδών ελευθεριών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και γι' αυτό θα πρέπει να τονίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα σύμπλεγμα αξιών και γι' αυτό έχουμε ενσωματώσει και τον χάρτη, τον χάρτη μελωδών δικαιωμάτων στην συνθήκη της Λισαβόνας, γι' αυτό έχουμε διοργανώσει πολλές ακροάσεις και έχουμε παραστεί σε πολλά φόρα και μας ενδιαφέρει να εξασφαλίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πλήρως προσιλωμένη σε αυτές τις αξίες και επίσης διότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ακούσει πολλές φορές κριτικές φωνές και επικρίσεις σε σχέση με τη στάση μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε τρίτες χώρες αλλά και σε σχέση με την ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς βρίσκεται, πώς, σε ποιο επίπεδο βρίσκεται η η διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τις διακηρύξεις μας, αλλά και σε σχέση με το άρθρο 2 της συνθήκης της Λισαβόνας. Έχουμε κάνει μια σειρά από ουσιαστικές συζητήσεις για τα θέματα αυτά στον χώρο της δικαιοσύνης, ελευθερίας και ασφάλειας, στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Είχαμε πολλές συζητήσεις, πολλές φορές έντονες και μέσα σε εισαγωγικά θερμές σε σχέση με τις συνταγματικές διασφαλίσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες. Ας δώσουμε λοιπόν τη δυνατότητα να ξεκινήσει η συζήτηση και απλώς θα σας πω ότι πρόσφατα τρεις από τις επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Επιτροπή Συνταγματικών Θεμάτων, η Νομική Επιτροπή και εμείς η Επιτροπή Δημοσίων Ελευθεριών έχουμε ε, εμπλακεί σε μια εσωτερική επαλεξέταση του προγράμματος της Στοκχόλμης για το χώρο ελευθερίας δικαιοσύνης και ασφάλειας βάσει του άρθρου 51 του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα πρέπει να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα, σε ποιο βαθμό έχουμε επιτύχει στην ε, σειρά των στόχων που είχαν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τις θεμελιώδες ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ποια είναι η ισορροπία που έχουμε επιτύχει, ποια είναι τα εκρεμή θέματα, πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την απόδοσή μας και να έχουμε μια καλύτερη υπο... ισορροπία μεταξύ ελευθερίας και ασφάλειας και πάνω απ' όλα πώς θα εξασφαλίσουμε ότι θα πλησιάσουμε τους πολίτες και κάποια θέματα πρόσφατα έχουν δημιουργήσει κάποιες ε, ανησυχίες. Οι αποκαλύψεις για το σύστημα PRISM παρακολούθησης των ε, Ευρωπαίων πολιτών από την Αμερικανική Υπηρεσία Ασφάλειας. Θα πρέπει λοιπόν να πλησιάσουμε τους Ευρωπαίους πολίτες και εν ώψη των εκλογών που επίκυνται το Μάιο του 2014, όπου οι, Ευρωπαϊκοί, οι πολίτες της Ευρώπης μάλλον θα έχουν τον αποφασιστικό ρόλο και για όλα αυτά είναι σημαντικό να θέσουμε στο επίκεντρο αυτής της συζήτησης και στο κέντρο της προεκλογικής εκστρατείας ανεξάρτητα από πολιτική παράταξη να κάνουμε σαφές ότι όχι μόνο έχουμε ασχοληθεί με την ε, χρηματοπιστωτική κρίση και τη διαχείριση του ευρώ, αλλά και με τις ελευθερίες και την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών και όταν διαπραγματευόμαστε και κάνουμε συμφωνίες εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτους, εξασφαλίσουμε ότι τα ευρωπαϊκά πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες και βρίσκονται σε όλα τα στάδια αυτής της διαδικασίας και ότι τηρούμε τα υπεσχημένα. Είναι λοιπόν πάρα πολύ θετική αυτή η άσκηση συνεργασίας μεταξύ της Υποπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, της Επιτροπής ε, ε, Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Δημοσίου Ελευθεριών και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι τμήμα αυτής της συζήτησης και θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Μόρτεν καταρχήν από τον Φορέα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Καλώς ήρθατε λοιπόν κύριε Κιέρουμ και σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κύριε, κύριε Πρόεδρε Φερνάνη. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να απευθυνθώ στις επιτροπές σας και να συνεχίσουμε τη συζήτηση που είχαμε ξεκινήσει πέρυσι τον Νοέμβριο για να συζητήσουμε την εσωτερική και εξωτερική διάσταση της συνοχής της πολιτικής δεν ανθρώπινα δικαιώματα. Χαίρομαι ακόμα περισσότερο που παρευρίσκονται και εκπρόσωποι των Εθνικών Κοινοβουλίων γιατί αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα να έχουμε μια πιο ευρεία συζήτηση και να έχουμε και την άποψη των κρατών μελών, να το δούμε το θέμα και από τις δύο του πτυχές των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμφωνώ με αυτό που ελέγχθη ότι για να είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση πιστική και να αποτελεί και πηγή έμπνευση για τους εταίρους μας στο εξωτερικό, πρέπει να, πρώτα απ' όλα να κοιτάξει τα του οίκου της, να δει πώς αντιμετωπίζει τις ε, προκλήσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο εσωτερικό της. Η συνοχή και η τήρηση των προτύπων ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν είναι απλώς μια ηθική υποχρέωση. Αυτές οι αξίες βρίσκονται στη βάση όλων των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε αυτές είναι ασκούνται στο εσωτερικό της, είτε προς το εξωτερικό. συχνά δεχόμαστε επισκέπτες από το εξωτερικό και ας μην είναι εντός της εντολής μου αυτό στην ε, Υπηρεσία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και διαπιστώνουμε ότι η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα μπορεί να εμπνεύσει συναδέλφους ή εταίρους σε άλλα μέρη του κόσμου. Όμως ταυτόχρονα γνωρίζουμε από τα στοιχεία που συγκεντρώνει η Υπηρεσία Θεμελιωδών δικαιωμάτων ότι υπάρχουν προβλήματα στην, στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διάφορα ζητήματα στα οποία θα επανέλθω. Αλλά μια γενική παρατήρηση που θέλω να κάνω από την αρχή είναι ότι το θέμα δεν είναι απλώς να έχουμε μια στιγμιαία εικόνα της κατάστασης ε, εδώ και τώρα των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Αυτό που έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι να εξετάσει κανείς εάν υπάρχει πρόοδος, εάν τα προβλήματα που εντοπίζονται αν... χάνουν αντιμετώπιση από τους θεσμούς, από την κοινωνία. Τελικά αυτό μας ενδιαφέρει και μας περισσότερο απ' όλα. Εάν υπάρχει αντιμετώπιση των προβλημάτων και των προκλήσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επομένω δεν μας ενδιαφέρει μόνο η εικόνα, μια φωτογραφία της σημερινής κατάστασης, αλλά επίσης να κοιτάξουμε και την ε, ε, πρόοδο και τη, τη συγκρίνουμε με προηγούμενες ε, καταστάσεις. Λοιπόν, πριν τώρα αναφερθώ στα κύρια ευρήματα της Υπηρεσίας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Θα ήθελα να τονίσω κάποια στοιχεία θετικά, κάποιους τομείς στους οποίους η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να συνεχίσει να ισχυρίζεται ότι είναι πρότυπο για άλλες περιοχές του κόσμου. Πρώτα απ' όλα σε καμιά άλλη περιοχή του κόσμου δεν υπάρχει τέτοιο υψηλό επίπεδο διαφάνειας όσον αφορά τη συζήτηση για το ποιες είναι οι προκλήσεις. Ε, υπάρχει ελευθερία του τύπου, υπάρχουν μέσα μαζικής ενημέρωσης τα οποία φωτίζουν αυτά τα ζητήματα ανθρωπινών δικαιωμάτων. Ταυτόχρονα υπάρχει ένα πολύ αποτελεσματικό και ενδελεχές ε, νομικό πλαίσιο. Η Χάρτα Ανθρωπινών Δικαιωμάτων που είναι νομικά δεσμευτική βρίσκεται στην κορυφή αυτή της πυραμίδας του νομοθετικού πλαισίου, αλλά επίσης έχει σημασία, έχουν σημασία και άλλες δράσεις, όπως για παράδειγμα η επικύρωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση της ε, Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Εκτός από αυτά τα νομοθετικά πρότυπα υπάρχουν και θεσμικά όργανα και σε εθνικό επίπεδο τα εθνικά δικαστήρια, αλλά επίσης και θεσμοί που εργάζονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα, η κοινωνία των πολιτών στα κράτη-μέλη, που φροντίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα να μην ξεχνιούνται ως θέμα, αλλά επίσης και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτή τη στιγμή η Χάρτα Ανθρώπινων Δικαιωμάτων υιοθετήθηκε, κυρώθηκε, το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή άρχισαν να ασχολούνται με αυτά τα θέματα πιο εστιασμένα, πιο εντελεχώς. και να αντιμετωπίζουν πλέον το ζήτημα της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, στο εσωτερικό των κρατών μελών. Επίσης υπάρχει μια σειρά συγκεκριμένων πολιτικών, για παράδειγμα για τους Ρωμά, για τους οποίους υπάρχει το Εθνικό ε, σχέδιο ε, ένταξης, ενσωμάτωσης. Οι πολιτικές επίσης έναντι ε, των θεγενών πληθυσμών και της καταπολέμησης των διακρίσεων. Οι επίσης οι πολιτικές μας για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, της, της σύγχρονης μορφής δουλεμπορίου ταυτόχρονα προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε πολύ σημαντικές προκλήσεις όσον αφορά την προστασία της προσωπικής ζωής και την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ένα θέμα επίκυρο. Ας μην ξεχνούμε λοιπόν αυτά τα βασικά θετικά στοιχεία που έχουμε στην Ευρώπη, στη διάθεσή μας. Όμως, όπω καλά γνωρίζουμε, άλλο πράγμα είναι νομοθεσία και άλλο πράγμα είναι η πρακτική εφαρμογή της. και θα ήθελα να δώσω ορισμένα παραδείγματα που έχουν σχέση επίσης και με την εξωτερική διάσταση. Φέτος, ο φορέας που προσωπώ, η Υπηρεσία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, έκανε μια έρευνα ε, ε, προσπαθώντας να χαρτογραφήσει την κατάσταση των δικαιωμάτων των ομοφιλοφίλων στα 27 κράτη-μέλη. Περίπου το 67% των απαντήσεων των ερωτώμενων μας απάντησαν ότι δεν ε, θα αισθάνονταν άνετα να κρατήσουν το χέρι του συντρόφου τους ε, σε δημόσιο χώρο που σημαίνει ότι ε, το πρόβλημα είναι υπαρκτό. Ακόμα περισσότερο να σκεφτούμε ότι το 1 τέταρτο των ερωτώντων μας είπαν ότι δέχτηκε βίαιες επιθέσεις τους τελευταίους 6 μήνες από την στιγμή που ε, διενεργήθηκε η έρευνα και όταν τους ρωτήσαμε τι, πώς αντέδρασαν, τι έκαναν για αυτό, απάντησαν ότι δεν απευθύνθηκαν στην αστυνομία γιατί δεν, δεν αισθάνονται ασφαλείς να απευθυνθούν στην αστυνομία ή θεωρούν ότι δεν θα κάνει τίποτα η αστυνομία. Επομένως η ΛΟΑΔ καλύπτονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, στο όσον αφορά τις διακρίσεις, την καταπολέμηση των διακρίσεων εναντίον τους, μόνο στον τομέα της εργασίας. Τον Ιούλιο του 2013 το Συμβούλιο υιοθέτησε της οδηγίε για την προώθηση και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των λεσβιών, ομοφιλοφίλων, αμφιφιλοφίλων και δεξουαλικών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να, ένα απτό παράδειγμα ε, όπου τα λόγια δεν συμβαδίζουν με την πράξη. Θα ήταν σκόπιμο ε, να υιοθετηθεί μια οριζόντια, μια γκάρσια ε, οδηγία καταπολέμησης των διακρίσεων, η οποία ανακαλύπτει όλες ε, τις ομάδες που υφίστανται διακρίσεις και όλους τους τομείς διάκρισης πέρα από τις διακρίσεις στην εργασία. Επίσης, θεμελιώδεις συνταγματικές αρχές ε, έχουν τεθεί στο στόχαστρο σε διάφορα μέρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως για παράδειγμα η ανεξαρτησία των δικαστηρίων, η ανεξαρτησία του συνηγόρου του πολίτη, και σε ορισμένες περιοχές ε, διαπιστώνουμε ατιμορουσία όσον αφορά τα εγκλήματα μίσους, δηλαδή τα εγκλήματα τα οποία στρέφονται κατά ε, ΛΟΑΔ, κατά εθνικών ή εθνοτικών μειονοτήτων. Και, ε, ενώ ταυτόχρονα αυτό είναι ένα από τα ζητήματα τα οποία ε, θέτουμε με το επιτάσσιο στις εξωτερικές μας σχέσεις. Το ζήτημα του ασύλου, της μετανάστευσης και της καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων, εδώ υπάρχει μια άμεση σχέση με την εξωτερική ε, διάσταση των πολιτικών μας, γιατί αναφερόμαστε πάντα σε επικόους τρίτων χωρών και σε διάλογο με τρίτες χώρες. Όπως θα γνωρίζετε προφανώς, χιλιάδες άνθρωποι πέθαναν προσπαθώντας να έρθουν στην Ευρώπη, στη Μεσόγειο. Χιλιάδες άνθρωποι πέφτουν θύματα εμπορίας ανθρώπων ε, και έρχονται στην Ευρώπη μέσω αυτών των κυκλωμάτων πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης, σεξουαλικής ή ε, εργάζονται υπό συνθήκες που προσυδειάζουν σε δουλεία. Αυτά είναι πράγματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε και θέματα που οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε. Υπάρχει νομοθεσία, υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο, αλλά δεν αρκεί αυτό. Πολλά θα μπορούσαν και θα έπρεπε να γίνουν. Χρειάζεται αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών ε, μελών της ε, Ένωσης στον τομέα του ασύλου και διαπιστώνουμε ότι αυτή η αλληλεγγύη είναι μάλλον περιορισμένη. Να σας δώσω ένα παράδειγμα οι Ηνωμένε Πολιτείε, για παράδειγμα, έχουν δεχτεί περισσότερες, περισσότερους πρόσφυγες από τη Μάλτα. Ναι. Θα μπορούσαμε λοιπόν να αναλάβουμε συγκεκριμένα βήματα. Και σε αυτή την προσπάθεια έχετε ρόλο να διαδραματίσετε εσείς ως μέλη των εθνικών σας κοινοβουλίων, σημαντικό ρόλο, να φροντίσετε αυτά τα θέματα να είναι στην ημερήσια διάταξη των κοινοβουλίων σας και να λαμβάνονται υπόψη ε, στην πράξη, στην καθημερινή πρακτική. Για παράδειγμα, τα Εθνικά Κοινοβούλια έχουν σημαντικό ε, ρόλο στη μεταγραφή του Ευρωπαϊκού Δικαίου στο Εθνικό Δίκαιο. Και άρα μπορείτε να εξασφαλίσετε κατά διάρκεια αυτής της μεταγραφής ότι οι θεμελιώδη δικαιώματα θα γίνονται σεβαστά στο Εθνικό Δίκαιο. Δεύτερον, η αποτελεσματικότητα αυτού του περίπλοκου μηχανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσε να βελτιωθεί με μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των επιτροπών που είναι αρμόδια για τα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα 28 κράτη-μέλη, αν υπήρχαν πιο συχνές συναντήσεις και πιο συχνά επικοινωνία για ανταλλαγή απόψεων και αναφέρομαι στις επιτροπές εκείνες που, και εκείνες που ε, ασχολούνται με εσωτερικά ζητήματα ανθρώπινων δικαιωμάτων και εκείνες που ασχολούνται με, την εξωτερική διάσταση. Τρίτο σημείο. Χρειάζεται συντονισμός, μεγαλύτερο συντονισμός σε εθνικό επίπεδο μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων στην προστασία και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. και τα εθνικά κοινοβούλια μπορούν να συμβάλλουν έτσι ώστε να υπάρχει συνεργασία και διάλογος μεταξύ όλων αυτών των φορέων. Τους φορείς αυτούς για την κοινωνία των πολιτών και να ανοίξω εδώ μια παρένθεση γιατί ένα από τα πράγματα που με απασχολούν είναι η αποδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών σήμερα στην Ευρώπη εν ώψη και ως αποτέλεσμα της ε, χρηματοπιστωτικής κρίσης. Η κοινωνία των πολιτών επλήγει ιδιαίτερα από την έλλειψη χρηματοδότησης και επίσης σε πολλές περιπτώσεις από την έλλειψη άλλων μορφών υποστήριξης. Και εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση όπως και τα κράτη-μέλη έχουν παίξει ένα ενεργό ρόλο για να υποστηρίξουν την κοινωνία των πολιτών και δεν πρέπει να παραμείνουμε μόνο στην κοινωνία των πολιτών έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά μας ενδιαφέρει και η δική μας κοινωνία των πολιτών που παίζει σημαντικό ρόλο στην προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε καθημερινό επίπεδο. Και τέλος, τονίζω ότι είναι απαραίτητο να συνεχίσουμε να συλλέγουμε περισσότερα και καλύτερα δεδομένα, ώστε να μπορέσουμε να αναπτύξουμε περιττέρω μια πολιτική ανθρωπινών δικαιωμάτων που να βασίζεται σε πραγματικά στοιχεία να μπορέσουμε λοιπόν να στοχεύσουμε καλύτερα τις πολιτικές μας και τους τρόπους παρέμβασής μας και φυσικά ο φορέας θεμελιωδών δικαιωμάτων είναι πάντα στη διάθεσή σας. <clears throat> σας ευχαριστώ λοιπόν για αυτή την ευκαιρία να παρουσιάσω τον φορέα μας. Ευχαριστώ κύριε Κέραμ και για τη δήλωσή σας και για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Βλέπω την πρότασή σας να συναντηθούν οι Επιτροπές Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε εθνικό επίπεδο και μετά το πρόβλημα είναι πώς μπορεί να συμμετάσχει και το ε, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν υπάρχει μια πλειοψηφία που να έχει υποστηρίξει μια, επιτροπή, μια πλήρης Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που να ασχολείται με τα εσωτερικά και τα εξωτερικά θέματα. Παραμένουμε λοιπόν ε, τμήμα της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και έχουμε κάποια δυνατότητα να επηρεάσουμε την λειτουργία της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ, αλλά δεν έχουμε ακόμα τον χαρακτήρα μιας Επιτροπής η οποία καλύπτει πλήρως και τον εσωτερικό και τον εξωτερικό χώρο. Είναι χρήσιμο όμως να βρισκόμαστε σε διαφορετικά επίπεδα και να συζητάμε μεταξύ μας ως Εθνικά και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και τώρα έχουμε τον ε, επικεφαλής της ομάδας του Συμβουλίου για τα θεμελιώδη δικαιώματα ε, και την ελεύθερη κυκλοφορία ατόμων, την κυρία Βιγκάντε Μίλια Σιούτε. Είναι η πρώτη φορά λοιπόν που έχουμε αυτή την ευκαιρία να ανταλλάξουμε αλλάξουμε μαζί σας, αν δεν κάνω λάθος. Χαίρομαι κυρία Πρόεδρε για την παρουσία μου εδώ και την ευκαιρία που μου δίνετε να κάνω μια σύντομη παρουσίαση. Το ΦΡΕΜΠ λοιπόν είναι το τμήμα που ασχολείται με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ελεύθερη διακίνηση των προσώπων. Είναι κάτι αρκετά πρόσφατο ακόμα αυτή η ομάδα εργασίας ακόμη ψάχνει την ταυτότητά της, ψάχνεται. Άρχισε ως ad hoc ε, ομάδα με κύριο καθήκον να διαχειριστεί την νομοθεσία στην οποία βασίστηκε το Ίδρυμα των Θεμελιωδών που ήταν και αυτή δικό μας έργο. Λοιπόν, από τότε που έγινε μια μόνιμη ομάδα εργασίας συνδεόμενη βέβαια με το Ίδρυμα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αλλά όχι μόνο. Τέθηκε ενισχύ και η συνθήκη της Λισαβόνας και η δουλειά μας καθορίστηκε από το κύριο γεγονός της συνυπογραφής από την ε, Ένωση της Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και μας πήρε πολύ χρόνο η προετοιμασία χωρίς να σημαίνει αυτό ότι μόνο αυτό κάναμε τόσο καιρό. Υπό την Ιρλανδική Προεδρία τον Ιούνιο του 2013 τα συμπαράσματα του Συμβουλίου για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα και την, ε, το κράτος δικαίου κατέληξαν στην έγκριση της συμπερίληψης της συνθήκη του, της Χάρτας των Θεμελιωδών και η συνυπογραφή α, της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θεωρήθηκε ως θεμελιώδες, θεμελιώδης πρόοδος για την πρόοδο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το συνδυασμό μεταξύ κράτους δικαίου και συγκεκριμένων θεμάτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ιδιαίτερα την καταπολέμηση της ξενοφοβίας, εγκλημάτων μίσους και της ομοφοβίας, ομοφιλοφοβίας. Στην την επόμενη προεδρία, το ΦΡΑΜΠ, η ομάδα εργασία μας δηλαδή, τόνισε κυρίως τέσσερα θέματα. Το πρώτο είναι η αποτελεσματικότητα της χρήσης των υπαρχόντων εργαλείων για την καταπολέμηση εγκλημάτων μίσους ή μισαλοδοξίας μάλλον και τουλάχιστον άρχισε μια συζήτηση για το τι θα έπρεπε ακόμη να επιτευχθεί στην Ένωση για την καλύτερη καταπολέμηση της μιχαλοδοξίας. Και ακούστηκαν πολλές ιδέες υπό την Ιρλανδική Προεδρία, ότι δηλαδή χρειάζεται προώθηση και του πολιτισμού ως ανθρωπίνο δικαίωμα, όχι μόνο νομοθεσία αλλά και ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζονται αυτά τα νομικά, οι νομικές ρήτρες και αν δεν ε, λειτουργούν καλά τι λείπει. Το σχέδιο της Προεδρίας ήταν πρώτον να συλλεχθούν πληροφορίες και δεδομένα για να μπορέσει να γίνει αυτή η συζήτηση. Ακόμη λοιπόν υπό την Ιρλανδική Προεδρία ζητήσαμε δεδομένα από το Ίδρυμα Θεμελιωδών και του ζητήσαμε να δει τα πράγματα από την άποψη των θυμάτων εγκλημάτων μίσους και μισολοδοξίας. Τι θα μπορούσε να γίνει για να προστατευτούν περισσότερο, μήπως χρειά, τα δικαιώματά τους, μήπως χρειάζεται και άλλη νομοθεσία ή τι άλλο. Εκτός αυτού, υπό τη Φιλανδική Προεδρία, Λιθουανική, ζητήσαμε στοιχεία για την καλύτερη καταπολέμηση της ξενοφοβίας μέσω νομοθεσίας. Ζητήσαμε συγκεκριμένα στο Συμβούλιο να ε, μας δώσουν τα κράτη-μέλη δεδομένα για την εμπειρία τους ως προς τη νομική συνεργασία σε αυτό το θέμα. Το ζητήσαμε και το κυριότερο είναι ότι οργανώνεται ετήσια κοινή συνεδρίαση Προεδρίας και Υπηρεσίας Θεμελιωδών για την καταπολέμηση της μυσαλλοδοξίας το ξαναλέω. Εδώ στις 13 Νοεμβρίου οργανώνεται, σας το διαφημίζω να το ξέρετε κι εσείς. Και ελπίζουμε να μας δοθεί εκεί η ευκαιρία να συζητήσουμε αληθινά πραγματικά προβλήματα και να ακουστούν εκεί καινούργιε ιδέε προ το τι θα μπορούσε να γίνει σε ευρωπαϊκό ενωσιακό επίπεδο για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Αυτό για την καταπολέμηση της μυσαλλοδοξία και των εγκλημάτων μίσου. Το επόμενο μας θέμα στο ΦΡΕΜΤ στην ομάδα εργασίας μας είναι το θέμα της εξωτερικής αποτίμησης, αξιολόγησης της υπηρεσίας θεμελιωδών. Σας το λέω καθαρά, δεν θα το κάνουμε εμείς πώς να το πω, δεν θα αξιολογήσουμε εμεί αυτή την υπηρεσία, έχει γίνει ήδη αξιολόγηση εξωτερικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο λοιπόν της υπηρεσίας διατύπωσε ορισμένες συστάσεις για το πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί η λειτουργία της, αν έπρεπε και πώς να αλλάξει ο σχετικός κανονισμός και στο Συμβούλιο σχεδιάζουμε την έγκριση των συμπερασμάτων του σχετικός όπου να εκφραστεί για ακριβώς αυτό το θέμα, τι πρέπει ακόμη να γίνει, τι λείπει για να γίνει πιο αποτελεσματική αυτή η υπηρεσία. Αλλά αυτό βέβαια είναι θέμα της Κομισιόν να υποβάλει καμία πρόταση που θεωρεί απαραίτητη. Τρίτο θέμα μας είναι τα δικαιώματα των ενωσιακών πολιτών και πιο συγκεκριμένα σχεδιάζουμε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για τα, ως προς τα συμπεράσματα της Κομισιόν για την ε, προστασία των πολιτών και των δικαιωμάτων τους. Τα συμπεράσματα θα ελπίζουμε να εγκριθούν τον Δεκέμβριο και να υποβληθούν στο Βίλνιους κατά τη λήξη της Προεδρίας. Πανηγυρική λήξη. Βέβαια δεν είναι δυνατόν να φανταστούμε, ε, θα ήταν δυνατόν να φανταστούμε την εργασία του Φρέμπτ αν δεν υπήρχε η υπογραφή της χάρτας, της σύμβασης. Μέχρι τώρα όμως οι συζητήσεις έγιναν άτυπα. Δεν έχει υποβληθεί ακόμα επίσημα η πρόταση. Πιο συγκεκριμένα τώρα για το θέμα εσωτερικής-εξωτερικής συνοχής. Στις 15 Σεπτεμβρίου εξετάσαμε ένα έγγραφο που θα γνωρίζετε κι εσείς που υπέγραψαν σα, καμιά σαρανταριά μη κυβερνητικέ οργανώσεις στο οποίο η κοινωνία των πολιτών εφιστά την προσοχή των ευρωπαϊκών θεσμών για το θέμα αυτό της σημασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των πολιτών και κάνει και ορισμένες συστάσεις για τη βελτίωση της κατάστασης, ειδικά δε συστάσεις προς εμάς. Εμείς το εξετάσαμε το έγγραφο και συμφωνήσαμε να το συζητήσουμε το Νοέμβριο την 1η μάλιστα Νοεμβρίου, ειδικά το θέμα δηλαδή της εξωτερικής εσωτερικής συνοχής και συνέπειας για τα ανθρωπίνα δικαιώματα και ο κύριος Σταύρος Λαμπρινίδης, ο πρόσωπος του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Υπηρεσίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα συνεννοηθούμε και προσπαθούμε να δούμε πώς θα μπορούσαμε καλύτερα να οργανωθούμε και να δούμε τι χρειάζεται να γίνει για να υπάρξει μεγαλύτερη συνέπεια ή συνοχή μεταξύ εξωτερικού και εξωτερικής διάσταση στα ανθρώπινα δικαιώματα. Και τώρα για να το συνδέσω με την πρωινή μας συζήτηση και τις δηλώσεις του πρεσβευτή του Συμβουλίου της Ευρώπης, προς το Συμβουλίο της Ευρώπης, θέλουμε να αποφευχθεί, να η πλημελής επιτήρηση ή εποπτεία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων χωρίς να υπάρχουν και επικαλύψεις. Και στο ΦΡΕΜΤ επίση συζητήσαμε σύντομα το θέμα της συνεργασίας μεταξύ Κομισιών και Συμβουλίου της Ευρώπης για να προετοιμαστεί το λεγόμενο Justice Scoreboard η, συνεργαζόμενη, συνεχιζόμενη συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης και την Κομισιόν υπάρχει, αλλά ταυτόχρονα ξέρουμε ότι χρειάζονται περαιτέρω συζητήσεις στο Συμβούλιο για να δούμε πώς τα στοιχεία του Συμβουλίου της Ευρώπης μπορούν να χρησιμοποιηθούν καλύτερα από, τους τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για τις ανάγκες της Ένωσης. Δέκα λεπτά μιλάω και θα μου ζητήσετε να σταματήσω φαντάζομαι σε λίγο. Γι' αυτό καταλήγω ότι για μας η συνέχεια της εργασίας του Συμβουλίου σχετικώς είναι πολύ σημαντική γιατί όπως ξέρετε υπάρχει εναλλασσόμενη προεδρία η κάθε μία βέβαια κληρονομεί ορισμένα θέματα στην άλλη αλλά για την καταπολέμηση της μυσαλλοδοξίας και των εγκλημάτων μίσους θα χρειαστεί να συνεχιστεί το πρόγραμμα και υπό την ελληνική προεδρία. Η συνέχεια λοιπόν είναι κάτι σημαντικό αλλά και η συνεργασία με εξωτερικούς αράγοντες. Εγώ είμαι ικανοποιημένη με τη συνεργασία που έχουμε με την υπηρεσία των θεμελιωδών, αλλά βέβαια υπάρχει χώρος και για βελτίωση. Και τώρα θα ακούσω δικέ σα ιδέε για τη βελτίωση των εργασιών μας. Σας κατευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Τασιούτε. Χαιρόμαστε επίσης για το γεγονός ότι έχετε και συζητήσεις για να εξασφαλίσετε το θέμα της συνακτικότητας των πολιτικών. Έχω τρεις ομιλητές από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Αν θέλετε να λάβετε το λόγο, παρακαλώ παρουσιάστε τον εαυτό σας. Ξεκινάμε από την κυρία Ροσάλια από τη Ρουμανία. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για όλους μας να μπορέσουμε να συζητήσουμε για τα θέματα αυτά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να πάρουμε και απτά παραδείγματα από την πρακτική που ακολουθείται σε άλλες χώρες και να ακούσουμε και τις απόψεις των άλλων κοινοβουλευτικών. Η Ρουμανία έχει ανακτήσει τη δημοκρατία πριν από 23 χρόνια και φυσικά εργαζόμαστε για να μπορέσουμε να επιτύχουμε μια συνεκτικότητα στην πολιτική μας στα εθνικά θέματα. Φυσικά έχουμε τεράστιες προκλήσεις σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα. και έχουμε καθυστερήσει πολλές φορές την ανάπτυξη της απαραίτητης νομοθεσίας. Συνεργαζόμαστε με την κοινωνία των πολιτών, αλλά υπάρχουν προβλήματα με την επίτευξη ίσων ευκαιριών από, για όλους λοιπά. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να δημιουργήσουμε αυτόν τον χώρο για τη στρατηγική που θέλουμε να εφαρμόσουμε και να κάνουμε και μια σωστή σχεδίαση των ε, ενεργειών μας. Είναι απαραίτητο πρώτα απ' όλα να έχουμε σχέδια δράσης τα οποία είναι ε, κατάλληλα για τις ιδιαιτερότητες κάθε κράτους μέλους και θα πρέπει να έχουμε και τις απαραίτητες μέρημνες για τη σωστή αξιολόγηση και τον έλεγχο όλων αυτών των ενεργειών. Οι νοοτροπίες αλλάζουν μόνο με πολύ βραδύ ρυθμό και γι' αυτό χρειαζόμαστε να έχουμε και μια υποστήριξη στις προσπαθίες μας. Δρούμε προς το συμφέρον όχι μόνο των πολιτών μας στη δική μας χώρα, αλλά και φυσικά προς το συμφέρον όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να κάνω και μια πρόταση. και χαίρομαι που αναφέρθηκε από τον κύριο <clears throat> κέρμε, για τη δημιουργία ενός ε, δικτύου εμπειρογνωμόνων που θα μπορούσαν να εργαστούν από κοινού για όλα αυτά τα θέματα. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να βρούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να μεταλαμπαδεύσουμε θετικές εμπειρίες από τα κράτη-μέλη μας, να έχουμε παραδείγματα με τα οποία θα βοηθήσουμε και τους ε, ομολόγους μας στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης να ε, εφαρμόσουν αυτές τις βέλτικες πρακτικές για την καλύτερη εφαρμογή των ε, θεμελιωδών ελευθεριών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτή είναι η πρότασή μου και ελπίζω ότι, μια, ότι οι συναντήσεις όπως η σημερινή θα συνεχίσουν να είναι πάρα πολύ σημαντικές για την εδραίωση ενός τέτοιου δικτύου και σε εθνικό αλλά και σε πανευρωπαϊκό δίκτυο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ακολουθεί η συνάδελφος από την Κροατία. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Μούλιτς. Άκουσα προσεκτικά τους ε, δύο προηγούμενους ομιλητές και οι δύο ανέφεραν ότι οι φορείς τους ε, εστίασαν ιδιαίτερα στα εγκλήματα μίσους και στην κατάρτιση κάποιων κατευθυντήριων οδηγών για την αντιμετώπιση της ε, μυσαλλοδοξίας και των εγκλημάτων μίσους. Εμείς το καλωσορίζουμε αυτό, το θεωρούμε εξαιρετική πρωτοβουλία ως μέλος του Κοινοβουλίου της ε, Κροατίας. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι προσπαθούμε και εμείς να φροντίσουμε το ποινικό δίκαιο στην Κροατία να προβλέπει ε, την δίωξη των ε, δραστών ε, εγκλημάτων μίσους, αλλά το ζήτημα είναι να, δούμε μάλλον και το ζήτημα της παρακίνησης σε εγκλήματα μίσους, το λεγόμενο hate speech, γιατί αυτό συνήθως προ υπάρχει των εγκλημάτων μίσους. Θα χρειάζεται ένα πλαίσιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο να ε, ενισχυθεί για την καταπολέμηση των διακρίσεων. Όσον αφορά την μεταχείριση των παράτυπων μεταναστών και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, πιστεύω ότι χρειάζεται να ενισχυθεί η συνεργασία με τρίτες χώρες αφενός και αφετέρου να ενισχυθεί η αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών. Χρειάζεται να βρούμε μια σωστή ισορροπία ε, και είμαι βέβαιος ότι οι συνάδελφοι από την Ελλάδα, από την Ιταλία, από τη Μάλτα καταλαβαίνουν πολύ καλά τι ε, εννοώ. Πολύ σύντομα η Κροατία θα γίνει το νέο κράτος μέλος που θα έχει την μεγαλύτερη ε, ε, τα μεγαλύτερα σύνορα στο εξωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επομένως είναι σημαντική η προστασία των εξωτερικών σύνορων, συμφωνούμε, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να φροντίζουμε για την δίκαιη και σύμφωνα με τα ανθρώπινα δικαιώματα μεταχείριση των παράτυπων μεταναστών. Πιστεύω ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και τα Εθνικά Κοινοβούλια θα κάνουν ό,τι μπορούν έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση τελικά να επικυρώσει τη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ελπίζω ότι η συνεργασία μας με το Συμβούλιο της Ευρώπης ε, θα συνεχίσει και θα ενισχυθεί μάλιστα. Πιστεύουμε ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης ε, και η τα πρότυπα, τα νομικά πρότυπα που έχει θεσπίσει είναι τα πλέον σημαντικά για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστούμε. Σε σχέση με το τελευταίο θέμα που αναφέρατε, υπάρχει μια ένα σχετικό ε, ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ζητά την κύρωση αυτή τη συνθήκη. Ε, αν θυμάμαι καλά πέρυσι το είχαμε συζητήσει έντονα. Ε, κάποια κράτη-μέλη επιθυμούν το αντίθετο δυστυχώς, προσπαθούν να καθυστερήσουν αυτή τη διαδικασία. Τώρα νομίζω βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο. Επίσης χρειάζεται οι υπηρεσίες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για παράδειγμα η Frontex, να έχουν ξεκάθαρη πολιτική όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, για παράδειγμα στον τομέα ε, της προστασίας των συνόρων. Και τώρα ένα συνάδελφος από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο κύριος Σταβάρης. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. <clears throat> Νομίζω ότι είναι μια θαυμάσια ευκαιρία για να συζητήσουμε θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων όσο, τόσο στο εσωτερικό και όσο και στο εξωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι που αφορά και εμάς τους ευρωβουλευτές όσο και τα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων. Έχουμε ένα νέο άρθρο στη Συνθήκη Λισαβόνα που αναφέρει ότι οι χώρες μας αποφάσισαν να δημιουργήσουν μία ένωση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1. Και το δεύτερο άρθρο αναφέρεται στους πυλώνες της ε, ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, σεβασμός για τα ανθρώπινα δικαιώματα, κράτους δικαίου, θεμελιώδε ελευθερίες κτλ. Όταν μιλάμε λοιπόν για τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτές είναι οι αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποφάσισαν τα κράτη-μέλη ότι θα είναι οι πυλώνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το τρίτο άρθρο που αναφέρεται στους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρεται ότι ο πρώτος στόχος είναι η ε, προώθηση αυτών των αξιών, η επίτευξη αυτών των αξιών και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πριν από την ενία αγορά, πριν από το Σέγγεν, πριν από οποιοδήποτε εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το 2012 ο στόχος Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η προώθηση και η εξασφάλιση των θεμελιωδών ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μας λείπει λοιπόν νομική βάση. Η νομική βάση υπάρχει, είναι πάρα πολύ σαφής. Απλώς πρέπει να υλοποιήσουμε αυτή τη νομική βάση με εργαλεία τα οποία πρέπει να διαμορφώσουμε από κοινού. Γι' αυτό είναι απαραίτητος ο διάλογος μεταξύ των ε, κοινοβουλίων και μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Παραγωγός χάρη η έκθεση της Κίνγκα Γκάλ το 2009 έχει μια σαφή πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να δημιουργηθεί ε, μια ομάδα εργασίας από, την, από το ομάδα εργασία ΦΡΕΜ του Συμβουλίου και την Επιτροπή Δημοσίων Ελευθεριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να κάνουν κοινέ συνεδριάσει σε τακτά διαστήματα. Υπάρχει λοιπόν αυτή η θέληση να προχωρήσουμε σε αυτήν την κοινή εργασία μαζί με το Συμβούλιο και με την Κομισιόν βέβαια. Μια άλλη πλευρά που είναι πάρα πολύ σημαντική είναι να μπορέσουμε να δώσουμε στον εαυτό μας τα απαραίτητα εργαλεία για να εξασφαλίσουμε ότι το κράτος δικαίου σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και επίπεδο κρατών ε, μελών δεν υποσκάπτεται από την οικονομική κρίση. Η ιστορία μας δείχνει ότι όταν υπάρχει μια οικονομική και κοινωνική κρίση αυτό οδηγεί σε μια κρίση του κράτους δικαίου και μια υποβάθμιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Αυτό λοιπόν μπορεί να μας φέρει αντιμέτωπους με προβλήματα που δεν ξέρουμε πώς θα τα αντιμετωπίσουμε. Σε μια πρόσφατη έκθεση για την οποία ήμουν υπεύθυνο, υπάρχουν προτάσεις για το πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε φορείς μη πολιτικού χαρακτήρα που θα επιτρέψουν να υποστηριχθεί το κράτο δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο φορέα θεμελιωδών ελευθεριών έχει ένα σημαντικό ρόλο, αλλά θα πρέπει να τροποποιήσουμε και το, την εντολή του φορέα θεμελιωδών δικαιωμάτων για να μπορέσει να εκφέρει γνώμη για θέματα τα οποία δεν είχαν τεθεί στην αρχή μέσα στην ε, σφαίρα εφαρμογής της, επειδή το Κοινοβούλιο είχε μια κάπως περιοριστική στάση. Επίσης, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι τα συντάγματά μας, οι δικαστικές μας αρχές, οι εισαγγελίες στα κράτη-μέλη μας θα δώσουν μια ιδιαίτερη προσοχή στα θέματα της ε, ισότητας των πολιτών και της μη παραβίασης των θεμελιωδών ελευθεριών. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχουν κατά κάποιο τρόπο επιτροπές Κοπενχάης μέσα εισαγωγικά για να εξασφαλίσουμε ότι σε κάθε μία από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι τηρούνται πάντα τα κριτήρια της Κοπενχάης. και αυτό θα πρέπει να εμπλέκει και την Επιτροπή η οποία θα πρέπει να τα εποπτεύει όλα αυτά. Πιστεύω ότι έχουμε το χρόνο ακόμα για να δημιουργήσουμε αυτό το οικοδόμημα, αλλά τα γεγονότα τα οποία βλέπουμε στις χώρες μας, η άνοδος του εξτρεμισμού, της πολιτικής βίας, οι πολιτικές δολοφονίες που είχαν πάψει να υπάρχουν στο ευρωπαϊκό έδαφος και επανέρχονται, όλα αυτά μας δείχνουν ότι ο χρόνος που έχουμε στη διάθεσή μας δεν είναι απεριόριστο και θα πρέπει το ταχύτερο δυνατό να μπορέσουμε να, να δράσουμε από κοινού για να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα θέματα, αλλιώς θα βρεθεί κάτω από μια τεράστια πίεση το κράτος δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ κύριε Ταβάρης. Πριν από τις στενές διακοπές εγκρίναμε την έκθεσή σας πράγμα. Και έχουμε και μια επιτροπή κοδονοκρουσίας κατά κάποιο τρόπο κινδύνου. Μια επιτροπή η οποία μπορεί να προειδοποιεί σε περιπτώσεις όπως αυτές που περιγράψετε. Ελπίζω ότι και στο μέλλον θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την επιτροπή και θα την κάνουμε να λειτουργήσει. ο κύριος Σωτήρχος από την Ελλάδα και μετά ο κύριος Καζάκ από τη Βουλγαρία. Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги. Наистина, първо, благодарности за организацията на тази... Σας ευχαριστώ πολύ ε, που διοργανώνετε αυτή την ε, συνάντηση με την εκπροσώπηση των μελών των Εθνικών Κοινοβουλίων και ε, την συμμετοχή των δύο επιτροπών ε, του Ευρωπαϊκού ε, Κοινοβουλίου. Γιατί πιστεύω ότι αυτό το ζήτημα, το ζήτημα της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι πάντα επίκαιρο. Ήταν στη βάση και στην θεμέλιο της ίδιας της ε, δημιουργίας ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρά το γεγονός ότι στην αρχή η Ευρωπαϊκή ε, Ένωση, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα ήταν μια οικονομική κοινότητα. Παρ' όλα αυτά, η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων Εναγράφει ήδη από τις ε, πρώτες θεμελιώδεις συνθήκες που δημιούργησαν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διανύσαμε έναν μεγάλο δρόμο ως Ευρωπαϊκή Ένωση ε, προασπίζοντας την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων κεφαλαίων αλλά και προασπίζοντας ε, θεμελιώδεις αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτές οι αρχές ε, βρίσκονται στη βάση της ε, ύπαρξης της Ευρώπης και ως Υπήρου ε, εδώ και αιώνες δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ήταν το λίκνο της δημοκρατίας πάντα αυτή η Ήπειρος. επομένως, χαιρετίζουμε τα βήματα που τα πιο πρόσφατα, για παράδειγμα την δημιουργία του φορέα θεμελιωδών δικαιωμάτων ή επίσης του εκπροσώπου για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Συνεχίζουμε με αυτόν τον τρόπο ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση να προασπίζει τα θεμελιώδη δικαιώματα με τον ίδιο τρόπο που προασπίζει την ελεύθερη οικονομία. Αλλά ας μην ξεχνάμε ότι πολύ σημαντικές προκλήσεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν και τα κράτη-μέλη και η Ένωση συνολικά. Και για να αντιμετωπιστούν αυτές τις προκλήσεις χρειάζεται συντονισμός και κοινέ πολιτικές συντονισμό σε όλα τα επίπεδα των θεσμικών οργάνων Και αυτό είναι απαραίτητο προκειμένου να γίνεται σεβαστή η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν εκφράζεται και όταν μιλά στην ε, παγκοσμίω στη διεθνή σκηνή. Θα ήταν λοιπόν ευκταίο όλα τα θεσμικά όργανα, όλοι οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μπορούσαν να έχουν μία φωνή για να εκφράζονται με μία φωνή όσον αφορά τις παραβιάσεις ανθρωπινών δικαιωμάτων και εντός και εκτός της Ένωσης. Πιστεύω πως σήμερα μία από τις πιο σημαντικές προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η Ευρώπη είναι το γεγονό ότι σε κάποιες χώρες που συνορεύουν με την Ένωση ε, έχουμε, ε, υπάρχει πόλεμος. Για παράδειγμα στη Συρία από την οποία πρόσφυγες πηγαίνουν προ την Τουρκία, προ την Κύπρο, προς την Ευρώπη και η αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, αυτών των καταστάσεων χρειάζεται μια ευρωπαϊκή πολιτική. Πρώτα απ' όλα πρέπει να συμφωνήσουν τα ίδια τα κράτη-μέλη, να εξασφαλίσουν αξιοπρεπείς συνθήκες σε αυτούς τους ανθρώπους. Συνθήκες στέγασης, διατροφής. Επομένως πρέπει να εκφραστεί ε, η αρχή της αλληλεγγύης. Για να μπορούμε να καταλήγουμε σε ενιαίες πολιτικές, οι οποίες τελικά να έχουν νόημα. Πολλά κράτη-μέλη επίσης αντιμετωπίζουν ε, προβλήματα με την κατάσταση των Ρωμά. Και εδώ είναι ένα τομέας στον οποίο απαιτείται αλληλεγγύη. Γιατί είναι ένα πρόβλημα κοινό, που το αντιμετωπίζουμε από κοινού δηλαδή, που ξεπερνά τα σύνορα των κρατών μελών και πρέπει να αντιμετωπιστεί επιγόντως. Πλησιάζουν οι εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Πολύ συχνά είμαστε έτοιμοι να προδώσουμε τις αρχές μας, να μην σεβόμαστε για παράδειγμα την αρχή της ισότητας, ε, προς άγραμ ψήφων. Η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και του Φορέα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα πρέπει να είναι σαφής και αυστηρή σε αυτόν τον τομέα. ότι η Μάλτα η κυρία Μπούτιτσεκ χαίρομαι πάρα πολύ που οι συνάδελφοι από τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρθηκαν σε προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν. Φυσικά ο καθένας αντιμετωπίζει τα προβλήματα από τη δική του πλευρά. Εγώ νομίζω ότι είναι τρία τα σημεία τα οποία θα ήθελα εγώ να τονίσω. Πρέπει να συνεργαστούμε πρώτα απ' όλα. τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι παραβιάσεις τους, ιδίως στις περιπτώσεις που συνδέονται με τη μετανάστευση, όλα αυτά δεν είναι προβλήματα μερικών μοναχα χωρών, είναι προβλήματα της σύνολης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δημιουργούν τα προβλήματα. Θα πρέπει να καταλάβουμε το, τη φύση του προβλήματος. Είναι το θέμα της αλληλεπίδρασης των πολιτισμών και των κοινοτήτων και φυσικά υπάρχουν διαφορετικές αντιμετωπίσεις από τη μια χώρα στην άλλη. Πρέπει να συνεργαστούμε, πάντα θέλαμε να προχωρήσουμε αυτήν την, ε, την διαδικτύωση μεταξύ μας. Συνεργαζόμαστε και με ΜΚΟ και είμαστε, θέλουμε να είμαστε πάντα κοντά στους ανθρώπους οι οποίοι υφίστανται δυσκολίες και βασάνους και φυσικά θα πρέπει να εργαστούμε και μαζί με όλους αυτούς τους πολίτες και να τους βοηθήσουμε γιατί είναι πολίτες οι οποίοι χρειάστηκε να φύγουν και να εγκαταλείψουν τις αιστείες τους. Δεν πρέπει να τους βλέπουμε σαν πρόβλημα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι μπορεί να είναι η λύση στο πρόβλημα που προσπαθούμε να λύσουμε. Ξέρουν ποια είναι τα προβλήματα στις χώρες τους, μπορούν να μας βοηθήσουν να καταλάβουμε καλύτερα πώς μπορούμε να συνεργαστούμε με τις χώρες τους, ώστε να μην υπάρξει αυτή η τεράστια πίεση στον πληθυσμό να φύγει. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι απλώς ένα όνειρο το οποίο σας παρουσιάζω. Πρέπει να εργαστούμε σκληρά προς την κατεύθυνση αυτή και να υποστηρίξουμε τις βασικές μας αρχές, τις αρχές της αλληλεγγύης και της αλληλοβοήθειας και νομίζω ότι όλοι και σαν άτομα και συλλογικά μπορούμε να προσφέρουμε το δικό μας πετραδάκι για τα θέματα αυτά. Το πρώτο πράγμα που έκανα όταν εξελεγήμουν στο Κοινοβούλιο της Μάλτας ήταν να προτείνω ένα νομοσχέδιο το οποίο ήθελε να υποστηρίξει την κοινότητα των ΛΟΑΔ και να αποτρέψει τις διακρίσεις εναντίον τους. Αυτές οι μικρές αλλαγές όμως σωρευτικά θα μπορέσουν να οδηγήσουν σε μεγάλες αλλαγές. Χαίρομαι που αναφερθήκατε στη Μάλτα, αναφέρθηκαν και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ιταλία όπως και η Ελλάδα, αλλά και πάλι δεν είναι μόνο τα δικά μας προβλήματα. Αυτά είναι προβλήματα τα οποία εμπλέκουν το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί, αλλιώς τα προβλήματα θα διωγγωθούν. Αν συνεργαστούμε όμως μπορούμε να βρούμε μια λύση, δεν έχω καμιά αμφιβολία. Η κυρία Φαρούτζια πάλι από τη Μάλτα. Εγώ Μαλτά. λέγομαι Φαρούτζια, είμαι από τη Μάλτα και όπως είπε και η συνάδελφός μου, θα ήθελα να υποθυμίσω σε όλους ότι επειδή η Μάλτα είναι τόσο μικρή χώρα και δεν έχει τόσο πολλούς πόρους και πολύ υψηλή πυκνότητα πληθυσμού, έχει ειδικέ ανάγκες. Ιδιαίτερες τουλάχιστον ανάγκες. Και όποτε τις αναφέρουμε χωρίς να αγνοούμε βέβαια την ανάγκη να υποδεχτούμε και πρόσφυγες, πάντοτε λέμε ότι δεν είμαστε σε θέση να δεχτούμε όλη αυτή την πίεση και όλους αυτούς τους πρόσφυγες όπως θα έπρεπε. Δυστυχώς οι Ηνωμένε Πολιτείε μόνο μας βοήθησαν μέχρι τώρα για να σηκώσουμε αυτό το βάρος και όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσπαθήστε να φανταστείτε τι εντύπωση δίνει αυτό σε άλλες υπήρους. Όταν βλέπουν δηλαδή ότι μια χώρα μέλος της Ένωσης έχει βοηθηθεί περισσότερο από χώρα εκτός της Ένωσης παρά από τις άλλες. Δεν νομίζω ότι αυτό δίνει καλή, δημιουργεί μια πολύ καλή εικόνα της Ένωσης προς τα έξω γιατί δίνουμε την εντύπωση ότι δεν βοηθάμε ο ένας τον άλλον και δεν μιλάμε με την ίδια φωνή. Οι αρχές της Ένωσης λοιπόν δεν γίνονται σεβαστές από τα ίδια της τα μέλη. Επαναλαμβάνω ότι είμαστε διατεθειμένοι να δεχτούμε όσο περισσότερους πρόσφυγες μπορούμε, αλλά χρειαζόμαστε γι' αυτό και τη βοήθεια άλλων χωρών. Ξέρουμε ότι και άλλες χώρες έχουν τέτοια παρόμοια προβλήματα αλλά πρέπει ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του και εμείς και οι άλλοι. Γι' αυτό σας υπενθυμίζω ακόμη μια φορά ότι οι πρόσφυγες αυτοί, οι παράνομοι αυτοί μετανάστες προσπαθούν να ξεφύγουν από τρομερές καταστάσεις στις χώρες προέλευσής τους και αυτό οφείλεται σε πολλά προβλήματα και καταχρήσεις και παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, τα οποία μπορεί να έχουν συμβάλει και χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει λοιπόν ως Ένωση στο σύνολό της να αντιμετωπίσουμε το ερώτημα κάνουμε ό,τι χρειάζεται και ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε τις αφρικανικές χώρες από όπου προέρχονται πολλοί από αυτούς τους πρόσφυγες. κάνουμε ό,τι μπορούμε ή μήπως περιοριζόμαστε στα λόγια ή πληρώνουμε μερικά χρήματα και θεωρούμε ότι κάναμε το καθήκον μας. Ξέρουμε ότι τέτοιου είδους χρήματα δεν φτάνουν πάντοτε σε αυτούς που τα χρειάζονται περισσότερο, στις χώρες προέλευσης δηλαδή. Και μαζί με τις άλλες χώρες που αντιμετωπίζουν τέτοιο πρόβλημα παράνομης μετανάστευσης, θα ήθελα να τονίσω ότι μακροπρόθεσμα πρέπει να δούμε το πρόβλημα στη ρίζα του και με τον πιο ρεαλιστικό τρόπο που θα μπορούσε να το λύσει για να υπάρξει περισσότερο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας για αυτούς τους ανθρώπους και να βοηθήσουμε και τις χώρες προέλευσής τους που βρίσκονται σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Ευχαριστώ με κοιτάξτε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ξαναγίνει συζήτηση πριν τις διακοπές για αυτό το θέμα και σκεφτήκαμε και εμείς πώς θα μπορούσε να γίνει πιο δεσμευτικό για όλες τις χώρες μέλη να πρέπει να δέχονται περισσότερους τέτοιους πρόσφυγες όπως στην Ελλάδα, Ιταλία, Μάλτα, Ισπανία. Δυστυχώς όμως οι περισσότεροι συνάδελφοι δεν δέχτηκαν την πρόταση αυτή, η πλειοψηφία δεν τη δέχτηκε να είναι νομικά δεσμευτικό. Πρέπει να το ξαναδούμε λοιπόν. Στην Επιτροπή Εξωτερικών οργανώσαμε πολλές ακροάσεις για να δούμε πώς θα μπορούσαμε να συνεννοηθούμε με χώρες του Μαγρέμπ ας πούμε γιατί ξέρουμε ότι πολλοί πρόσφυγες έρχονται, ξεφεύγουν από σειράξεις όπως στο Ιράκ ή στην Υποξαχάρια Αφρική και όταν κλείνουν τα σύνορα δεν μπορούν πια να φύγουν από πουθενά. Οι περισσότερες χώρες βέβαια προβλέπουν διαδικασίες για τη χορήγηση ασύλου αλλά η Επιτροπή Εξωτερικών και η δική μου Επιτροπή και η ΛΥΜΠΕ σίγουρα έχει συζητηθεί πολλές φορές, μπορώ να σας διαβεβαιώσω και εμείς ως πολιτικοί εδώ, που εκπροσωπούμε τις χώρες μας δεν θέλουμε να θανατώνται, να πεθαίνουν τόσες χιλιάδες άνθρωποι κάθε χρόνο στα εξωτερικά μας σύνορα. Πρέπει να βρούμε μια πολιτική λύση. Και τώρα έληξε ο κατάλογος, εξαντλήθηκε ο κατάλογος ομιλητών από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Αν θέλει κανείς να μιλήσει να μου το πει τώρα και οι ευρωβουλευτέ ούτε. Τότε θα δώσω το λόγο στο δίκτυο ΜΚΟ ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η κυρία ούτε το ανέφερε και πριν. Πέστε μας και εσείς τι θα μπορούσε να κάνει το Συμβούλιο για να αντιμετωπίσει καλύτερα και συνεπέστερα το πρόβλημα. Χαίρομαι για την παρουσία σας. Είστε ο κύριος Νίκολα Βέγκερ, η κυρία. Ας ακούμε. Ο κύριος. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και κύριε Λόπες Αγγελάρ για την ευκαιρία μας δίνετε. Λέγομαι Νίκολα Βέγγερ και εκπροσωπώ όπως είπατε το δίκτυο κοιό ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το είπε και η κυρία προηγουμένως ασχολούμαστε κυρίως με θέματα εξωτερικών σχέσεων, αλλά τελευταία και για το θέμα της συνοχής συνέπειας νεκτικότητας εσωτερικών εξωτερικών. Οι ΜΚΟ τεκμηριώνουν σταθερά δεδομένα για τα προβλήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά είμαστε πολύ μακριά από τις δηλώσεις της Λέδης Άστον για το Silver Thread των εξωτερικών σχέσεων και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν έχει ακόμα τίποτα πλήρως εφαρμοστεί. Παρακαλώ λίγο πιο αργά, λίγο πιο ήσυχα, γιατί δεν μπορούμε να καταλάβουμε η <laughs> μεν δε αυτό Ορίστε κύριε μου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εφαρμογή της χάρτας δεν πέτυχε πλήρη εφαρμογή. Οι διαδικασίες για παραβίαση των ορισμένων ε, χωρών μελών δεν έχουν καταλήξει και οι αποφάσεις λαμβάνονται με διαφανή τρόπο και πολλές φορές γίνονται διακοσμητικές μόνο αλλαγές. Η ετήσια έκθεση της Κομισιόν για τη Χάρτα δεν αναφέρει όλα τα στοιχεία ενώ τα έχει. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει μιλήσει καμιά φορά λίγο πιο θαραλέα, όπως ας πούμε για την Ουγγαρία και για τις εκθέσεις για τις επανεισδοχές. Αλλά φυσικά επηρεάζεται από την κυριαρχούσα πολιτική κατάσταση και γι' αυτό η τελευταία του έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν ανέφερε, δεν έκανε καμία επίκριση για καμία χώρα συγκεκριμένα. Εδώ πρόκειται όμως για σοβαρές παραβιάσεις των αρχών και δικαιωμάτων που εγκρίνει η Ένωση και μόνο οποίοι βλέπουμε. Τα τελευταία συμπεράσματα του Συμβουλίου αναφέρουν την πιθανή ανάγκη η εξέβρεση μιας μεθόδου αντιμετώπισης των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά στο State of the Union ο πρόεδρος Μπαρόσο δεν έδωσε καμία απάντηση στα κυριότερα προβλήματα που έχουμε ταυτίσει. Είναι λοιπόν σημαντικό νομίζουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μαζί με τα εθνικά πρέπει να συνεχίσει να προωθεί ενεργά την ανάγκη να υπάρξει συντονισμό τη πολιτική για θέματα βαρβία ανθρωπίνων δικαιωμάτων με συγκεκριμένε προτάσει και παραδείγματα. Καλούμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά να το πράξουν αυτό. Πρέπει να υπάρξει και ένα περαιτέρω έγγραφο εκτός από το σχέδιο πλαίσιο που το δεχόμαστε φυσικά. Όλα τα κράτη-μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο, του Συμβούλιο πρέπει από κοινού να εφαρμόσουν ένα πρόγραμμα πλαίσιο που να χρησιμοποιεί όλα τα διαθέσιμα εργαλεία που διαθέτει. Τίποτα λιγότερο δεν πρόκειται να έχει αποτέλεσμα. Εκτός από μια στρατηγική πλαίσιο δηλαδή, θα μπορούσαν να γίνουν ήδη από τώρα και ορισμένα συγκεκριμένα πράγματα. Πρώτον, χρειάζεται, πρέπει το ΦΡΕΜΠ να έχει μια πιο θαραλέα εντολή. Να, δοθεί, να δίνεται μια επίσημη απάντηση από το Συμβούλιο για τις σχετικές εκθέσεις του Κοινοβουλίου και του ΦΡΕΜΠ. Και να υπάρχει μεγαλύτερη συνεργασία και με το Συμβούλιο της Ευρώπης και της ΜΚΙ γιατί ξέρουμε μερικές όπως τη δική μου που δεν έχουν κληθεί ποτέ. Δεύτερον, χρειάζεται συγκεκριμένο και λεπτομέρειες σχέδιο από την Κομισιόν για τις διαδικασίες για παραβίαση, για παράληψη. Έχουν ληφθεί μεν ορισμένα μέτρα εξακρίβωσης, αλλά χρειάζεται περισσότερη διαφάνεια όλα αυτά. Αλλά θα να γίνει μια νέα δήλωση σχετικά με το άρθρο 7 και μία πιο αποτελεσματική στρατηγική για την εφαρμογή της χάρτας των θεμελιωδών που θα επέτρεπε μια σωστή αξιολόγηση και υποπτία. Πιστεύουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έπρεπε να κάνει συγκεκριμένε συστάσει στα κράτη-μέλη όπου τα θέματα της παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων να έχουν εξακριβωθεί. Και τέλος, ενθαρρύνουμε όλους εδώ μέσα να ζητήσουν στεναρότερη εντολή για την υπηρεσία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αναφέροντας συγκεκριμένα τα άρθρα 2 και 7. Δεν είναι εύκολο πράγμα, αλλά νομίζουμε ότι είναι κάτι απαραίτητο και βιώσιμο. Τα εργαλεία υπάρχουν, παραμένει θέμα πολιτικής θέλησης και οράματος. Η Ένωση έχει καταφέρει να δημιουργήσει μία στρατηγική για τα ανθρώπινα δικαιώματα και είμαι πεπισμένο εξωτερικά και είμαι πεπισμένο ότι μπορεί να το κάνει και για τα εσωτερικά. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Ευχαριστώ Νικολά. Αναφέρθηκε στο Κοινοβούλιο και στη δράση του ΦΡΕΜΤ η κυρία Μισελίτη. Πρέπει να φύγει όμως, θα της δώσω πρώτα τον λόγο για να απαντήσει και μετά μπορούμε να συνεχίσουμε. Σας ευχαριστώ για αυτές τις θετικές προτάσεις. Βέβαια, τις έχω ξανακούσει και στο παρελθόν. Η συζήτηση που προετοιμάσουμε για τις 21 Νοεμβρίου θα είναι ένα πρώτο βήμα στην σκέψη μας για το πώς μπορούμε να αναπτύξουμε καλύτερα τις ενέργειές μας στον τομέα αυτό. Είναι η πρώτη, το πρώτο στάδιο για να υπάρξει ένας πιο ανοιχτός χαρακτήρας στο ΦΡΕΜΠ e και πιστεύω ότι αυτό μπορεί να γίνει με βαθμίο τρόπο. Δεν μπορώ να σας υποσχεθώ ότι θα καλέσουμε αμέσως εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών σε αυτήν την ομάδα εργασία. Αλλά καταγράφω αυτά που είπατε και θα μεταφέρω και το μήνυμα αυτό στους συναδέλφους μου στην ΦΡΕΜΠ. Η δική μας άποψη είναι ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε αποτελεσματικούς τρόπους συνεργασίας με εξωτερικούς φορείς και ένα από τα θέματα που πρέπει να σκεφτούμε είναι το, η έκταση της κοινωνίας των πολιτών και ο αριθμός των φορέων που θα θέλουμε να ε, έχουμε να συνεργαστούμε μαζί. Είναι ένα από τα θέματα, δεν ξέρω αν σας ικανοποιούν αυτά, αλλά αυτά μπορούσα να σας πω τώρα. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Και νομίζω θα ξαναγυρίσετε στην Βίλνιους τώρα. Όπως ε, και το πρωί έχουμε ενώπιόν μας τον εκπρόσωπο από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ιδρυμάτων για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Ίσως θέλετε να λάβετε το λόγο και εσείς να πείτε κάτι. Η εξωτερική διάσταση της ελευθερίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι ένα θέμα πολύ ευρύ. Γι' αυτό εγώ θα εστιαστώ μόνο σε ορισμένες πτυχές που θεωρώ ε, μεγάλη σημασία. Πρώτα απ' όλα το στρατηγικό σχέδιο και το σχέδιο δράσης του 2012 είναι ημιτελές, είναι ανεπαρκές γιατί αναφέρεται μόνο σε ορισμένα θέματα. Η ετήσια έκθεση του 2013 είναι ακόμα μικρότερη και αναφέρεται ουσιαστικά μόνο σε ένα θέμα την εμπορία ανθρώπων. Ευελπιστώ η Ευρωπαϊκή Ένωση τα επόμενα χρόνια να καταφέρει να υιοθετήσει ένα πιο συνεκτικό, πιο πλήρες πρόγραμμα ανθρωπινών δικαιωμάτων και να καλύψει και άλλα σημαντικά θέματα, τα οποία ε, για να αντιμετωπιστούν θα πρέπει η στρατηγική να έχει σαφείς στόχους και θα φέρω ένα παράδειγμα. Το παράδειγμα της ε, Ρουμανίας, εκεί θα μπορούσαν να τεθούν συγκεκριμένοι στόχοι ε, όσον αφορά το, τη διαφάνεια. Είναι προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και των κρατών μελών της η στρατηγική για την αναπτυξιακή συνεργασία να ευθυγραμμιστεί με τα προγράμματα ανθρωπινών δικαιωμάτων έτσι ώστε να υπάρξει αντίκτυπος ε, επιτόπου. Αυτή η παγκόσμια πρόκληση των ανθρωπινών δικαιωμάτων πρέπει να ε, τη λάβουμε υπόψη μας σοβαρά και όταν σχεδιάζουμε πολιτικές ανθρωπιστικής βοήθειας και αναπτυξιακής συνεργασίας. Εκεί είναι ένας τομέας πολιτικής όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να επηρεάσει τα πράγματα. Αναφέρθηκα σε μια πιο έξυπνη στρατηγική ε, για την αναπτυξιακή συνεργασία. Για να ενσωματωθεί μια διάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε αυτές τις πολιτικές, χρειάζεται σχεδιασμός και επίσης ε, να επιλεγούν με τρόπο ε, διαφανή τα ζητήματα στα οποία θα εστιάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποτέ κανείς δεν μπορεί να αντιμετωπίζει όλα τα θέματα, επομένως θα πρέπει να επιλέξει η Ευρωπαϊκή Ένωση ορισμένα και αυτό πρέπει να γίνει με τρόπο διαφανή. ευελπιστώ ότι το στρατηγικό πλαίσιο θα μπορέσει να βελτιωθεί και να αποκτήσει στρατηγικούς στόχους και προτεραιότητες. Και τέταρτον, προηγουμένως ανέφερα ότι στα περισσότερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπάρχουν ανεξάρτητες επιτροπές ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εθνικές επιτροπές αυτές οι Εθνικές Επιτροπές Ανθρωπινών Δικαιωμάτων μπορούν να συμβάλλουν και στην εσωτερική αλλά και στην εξωτερική διάσταση. Αυτές οι Επιτροπές Ανθρωπινών Δικαιωμάτων συνεργάζονται ε, επίσης ε, και με άλλους φορείς για την εκπαίδευση, δημιουργούν δίκτυα. Έχουμε δημιουργήσει μια Διεθνή ε, Επιτροπή Συντονισμού των Επιτροπών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην οποία πρόεδρος πολλά χρόνια ήταν ο προκάτοχός μου. Σε, αυτή την, σε αυτόν τον φορέα συμμετέχουν επιτροπές από την Αφρική, από την Ασία, οι οποίες πολλές φορές ε, μπορούν να φροντίσουν για τη λογοδοσία των υπετίων στις χώρες τους πολύ καλύτερα από ότι εμείς. αλλά θα πρέπει να δημιουργηθούν εθνικές επιτροπές ανθρωπινών δικαιωμάτων σε όλα τα κρατη και να ενισχυθούν οι ήδη υφιστάμενες. Πολύ συχνά αυτές οι εθνικές επιτροπές δεν έχουν τους οικονομικούς πόρους και τους ανθρώπινους πόρους που χρειάζονται για να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία τους και να επιτελούν το καθήκον τους. Και πέμπτον, ένα θέμα που έχω αναφέρει πολλές φορές και κατά το παρελθόν, θα πρέπει να γίνει μία ανεξάρτητη αξιολόγηση της, νομο... της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στο μέλλον. Ίσως αυτό θα μπορούσε να το αναλάβει ο Φορέας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Πιστεύω ότι αυτό είναι ίσως μια ιδέα που θα έπρεπε να εξετάσουμε. Πέρα λοιπόν από αυτές τις συστάσεις που ήδη έκανα, οι προτάσεις μου θα ήταν οι εξής. Θα πρέπει να μας προβληματίσει το γεγονός ότι το στρατηγικό σχέδιο και το ε, πρόγραμμα δράσης του 2012 και 2013 δεν είχαν ε, επαρκές εύρος και επίσης δεν είχαν προτεραιότητες και στόχους. Όπως προανέφερα θα πρέπει να ενισχυθούν οι Εθνικές Επιτροπές Ανθρωπινών Δικαιωμάτων όχι μόνο στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και σε ολόκληρο τον υπόλοιπο κόσμο για να μπορούν αυτές οι Εθνικές Επιτροπές Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να λειτουργούν με ανεξαρτησία και ε, με επάρκεια, χρειάζονται ε, τη συμβολή, ε, χρειάζονται πόρους και επίσης ένα πολιτικό πλαίσιο. Και στις περιοχές όπου ήδη υπάρχουν τέτοιες επιτροπές, αυτές θα μπορούσαν να ενισχυθούν. Ευχαριστούμε. Thank you, Madam, Madam Chair. Uh, I will continue in Polish language. Πολωνικά θα συνεχίσω. Ευχαριστώ. Έχω παρακολουθήσει με μεγάλο ενδιαφέρον την συζήτηση αυτή και ιδίως αυτά που είπε ο προλαλής σας. είναι πολύ σημαντικό το ότι ως εκπρόσωπος μια μης μη κυβερνητική οργάνωση κρίνει αυτά τα οποία προσπαθούμε να κάνουμε εμεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Η σχέση μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των κυνηγών και, των, συγγνώμη, και της κοινωνίας των πολιτών παίζει ένα ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο. Έχω προσπαθήσει μέσα στην Επιτροπή και την υποεπιτροπή μας θα έχω προσπαθήσει ε, να, επιτύχω συνειδητοποίηση των συναδέλφων μας περισσότερο σε σχέση με το τι μπορούν να κάνουν οι εθνικοί φορείς και τα εθνικά ιδρύματα και πώς μπορούμε ιδιαίτερα να χρησιμοποιήσουμε αυτούς τους φορείς για μια πιο στενή εταιρική σχέση με, τους, με τις γειτονικέ μας χώρες. Παραδείγματος χάρη, τα θέματα της συνεργασίας των διοικητικών επιτρόπων των Ombudsman με τις γειτονικέ χώρες. Αυτό είναι μια πρωτοβουλία η οποία ξεκίνησε από τον Πολωνό διαμεσολαβητή, η Διοικητικό Επίτροπο, ο οποίος ξεκίνησε <clears throat> μια συνεργασία με τον ομόλογό του στη Γαλλία. Η προσπάθεια ήταν να αλλάξουμε την μορφή της συνεργασίας μας με τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, αλλά να δείξουμε πως μια χώρα όπως η Πολωνία που ήταν τότε μέσα σε μια διαδικασία πολιτικής μετάβασης αντιμετωπίζει θέματα όπως αυτά της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν είναι λοιπόν μονάχα για συναντήσεις και συζητήσεις, αλλά και πρακτικές αλλαγές, ανταλλαγές απόψεων για συγκεκριμένα θέματα. Ο στόχος μας ήταν να δούμε πώς στο σύνολο αυτό της διαδικασίας στην Πολωνία μπορούμε να δώσουμε απάντηση σε συγκεκριμένα ερωτήματα. Παραδείγματος χάρη, η κατάσταση των γυναικών στις <clears throat> φυλακές ή επίσης <clears throat> θέματα όπως το εργασιακό δίκαιο και η εξασφάλιση μιας ισορροπίας μεταξύ εργοδοτών και εργασομένων επίσης η αντιμετώπιση των διακρίσεων στον χώρο εργασίας, αλλά όχι μόνο εκεί, και επίσης το θέμα της προστασίας της νεότητος των παιδιών και των νέων. Υπήρξε λοιπόν μια πολύ ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων μεταξύ διαμεσολαβητών. Και οι εκπρόσωποι των κρατών μελών, καθώς και οι εταίροι μας, έχουν προσπαθήσει να δείξουν ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλες οι χώρες είναι παρόμοια. Αυτό έκανε ιδιαίτερα καρποφόρα την ανταλλαγή απόψεων. Προφανώς δεν είχαν όλη τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε αυτή την διαδικασία ανταλλαγής απόψεων και επομένως δεν είχαμε γενικά τη δυνατότητα να συμμετάσχουν όλοι σε αυτή την εταιρική σχέση. Πιστεύω όμως ότι παρόλα αυτά είναι απαραίτητο να τονίσουμε ότι οι εθνικοί φορείς που ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν ένα μεγάλο απόθεμα γνώσεων και εμπειριών. Υπάρχουν καλά παραδείγματα, υπάρχουν και κακά παραδείγματα, καλές και κακές εμπειρίες, αλλά μέσα από αυτή τη διαδικασία μπορούμε να επιλέξουμε τις βέλτιστες πρακτικές που μπορούν να μας επιτρέψουν να πετύχουμε τους στόχους μας και συγκεκριμένα καταδείξαμε πως χώρες που βρίσκονται σε μετάβαση μπορούν να πράξουν τα απαραίτητα για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επίσης υπάρχουν προβλήματα σε σχέση με την εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Υπήρξε μια επιφυλακτική στάση από πολλούς εναντί της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί θεωρήσανε μερικοί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί με το στανιό να εφαρμόσει ορισμένες ε, ε, διαδικασίες. Θα πρέπει πάντα να αφήσουμε τους ανθρώπους να αντιμετωπίσουν αυτά τα πράγματα βάσει των δικών τους πολιτιστικών παραδόσεων και μέσα στην οτροπία Του Ένα δεύτερο στοιχείο είναι ότι προσπαθήσαμε μέσα στην ε, υποεπιτροπή μας να αντιμετωπίσουμε το εξής θέμα. Ένα θέμα το οποίο και τώρα μας απασχολεί. Πρόκειται για την εταιρική ευθύνη των ε, επιχειρήσεων. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι ε, επίκαιρο σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλες οι χώρες αυτές και ακόμα και ο ΙΕ πρέπει να αντιμετωπίσουν και να επιληθούν το θέμα αυτό. Του θέματος αυτού βέβαια υπάρχουν διαφορετικές ε, παραδόσεις σε, από κράτος σε κράτος. Τα σκανδιναβικά κράτη έχουν ήδη δώσει την πρέπουσα σημασία σε όλα αυτά τα θέματα και εγώ πιστεύω δεν υπάρχει λοιπόν έλλειψη θεμάτων που μπορούμε να συζητήσουμε μαζί με τους εταίρους μας στην Ανατολική Ευρώπη και μαζί με την κυρία Γκόμες έχουμε μιλήσει και για το Πακιστάν και για τα θέματα της παιδικής εργασίας εκεί. Υπάρχει φυσικά μια εμπορική, εμπορικού, υπάρχουν εμπορικού χαρακτήρα συμφωνίες με πολλές χώρες του κόσμου όπου υπάρχει παιδική εργασία. <clears throat> Είναι χώρες όπου υπάρχει εκμετάλλευση της παιδικής εργασίας και τα προϊόντα που προέρχονται από αυτή την εκμετάλλευση της παιδικής εργασίας εξάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γνωρίζουμε όλοι τι συνέβη στο Μπαγκλαντές, όπου εργαζόντουσαν άνθρωποι κάτω από σκανδαλώδεις συνδίκες και έχασαν και τη ζωή τους στη συνέχεια. Όλα αυτά μας οδήγησαν στο να ζήσουμε μια τεράστια τραγωδία. Αυτό σημαίνει ότι σε πάρα πολλού τομεί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπάρχουν οι δυνατότητε να καταλήξουμε σε μια κοινή κατανόηση και πιστεύω ότι η εταιρική ευθύνη των επιχειρήσεων, η εργασία των παιδιών, η εργασία των γυναικών, όλα αυτά που έχουν να κάνουν με την εκμετάλλευση των εργαζομένων, θα παίξουν και ένα ακόμα μεγαλύτερο ρόλο στο μέλλον και γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει εμεί να πάρουμε αυτή την πρωτοβουλία, να προχωρήσουμε και να εξασφαλίσουμε μια καλύτερη συνεργασία στα θέματα αυτά. Ευχαριστώ κύριε Τσίπ και ξαναγυρίζω σε ορισμένα από τα ερωτήματα τα οποία τέθηκαν. Δίνω το λόγο στον εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Φορέα για τις θεμελιώδεις ελευθερίες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σχολιάσω ορισμένα από αυτά που ακούστηκαν. Πρώτα απ' όλα η κυρία Μπύρο από Ρουμανία αναφέρθηκε στο ζήτημα των εθνικών στρατηγικών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τι είδου υποστήριξη θα μπορούσε να δοθεί και τι συνεργασία θα μπορούσε να υπάρξει μεταξύ των κρατομελών στην κατάπτυση και υλοποίηση αυτών των στρατηγικών. Θα ήθελα να σας δώσω ένα παράδειγμα από κάτι που ήδη συμβαίνει. Όταν, έγινε, δημοσιεύθηκε η ανακοίνωση για τους Ρωμά, το 2011 από την Επιτροπή, ένα σημαντικό στοιχείο αυτής της ανακοίνωση ήταν ε, ε, η αναφορά που έλεγε ότι θα έπρεπε να υιοθετηθούν από τα κράτη-μέλη εθνικές στρατηγικές ενσωμάτωσης των Ρωμά. Και τότε ζητήθηκε από το Φορέα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων να βοηθήσει τα κράτη-μέλη στην ανάπτυξη αυτών των στρατηγικών η ανάπτυξη των στρατηγικών έγινε από τα κράτη-μέλη στη συνεργασία με την Επιτροπή, αλλά η Φορέα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων συνέβαλε και επίση κυρίω ε, αυτό στο οποίο δραστηριοποιήθηκε ο φορέα ήταν η παρακολούθηση τη υλοποίηση αυτών των στρατηγικών. Τι είδου δείκτε μπορούμε να αξιοποιήσουμε για να δούμε εάν αυτέ οι στρατηγικές υλοποιούνται. Ε, έχουν αναλυφθεί νομοθετικές πρωτοβουλίες, έχουν ε, γίνει βήματα ε, για την ενσωμάτωση αυτής της συγκεκριμένης περιθωριοποιημένης ομάδας. Ένα παράδειγμα λοιπόν συνεργασίας. Πολλά κράτη-μέλη συμπεριλαμβανομένες και της Ρουμανίας συνεργάστηκαν σε αυτήν την διαδικασία και νομίζω ότι αντλήσαμε διδάγματα και φάνηκε ποιο ε, θα μπορούσε να είναι ο ρόλος του Φορέα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στην ανταλλαγή πληροφοριών και στην διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών. Αυτή λοιπόν η ανταλλαγή απόψεων την οποία διαπιστώνω κάθε φορά που επισκέπτω με ένα κράτος μέλος. Ε, συζητάμε με τους υπουργούς ε, δικαιοσύνης, παιδείας, και μου αναφέρουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, πάντα εγώ τους ρωτώ, ε, δεν απευθύνεστε σε ομολόγους σας, σε άλλα κρατημέλη, δεν συζητάτε τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε αφού είναι κοινά εξάλλου. Ε, διαπιστώνω ότι όχι, δεν υπάρχει αυτή η συνεργασία. Ε, ο Φορέας Ανθρωπινών Δικαιωμάτων έχει περιορισμένους πόρους στη διαθεσή του, αλλά σίγουρα θα μπορούσε, ακολουθώντας το παράδειγμα της στρατηγικής για τους Ρωμά, να διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Και τώρα ε, έρχομαι σε αυτό που είπε η κυρία Μιούλεκ από την, Κροα... Μούλιτς, από την Κροατία. Αναφερθήκατε στο ρόλο του Συμβουλίου της Ευρώπης. Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί η συνεργασία, η αλληλεπίδραση ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα του Φορέα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, φαινός και αφετέρου του Συμβουλίου Ανθρωπινών Δικαιωμάτων. Φυσικά ε, δεν είναι μυστικό ότι όταν δημιουργήθηκε ο Φορέας Ανθρωπινών Δικαιωμάτων το Συμβούλιο της Ευρώπης ήταν κάπως ανήσυχο μήπως ε, μπούμε στα χωράφια του τροποντινά αλλά νομίζω ότι αυτή η συζήτηση για την αλληλοεπικάλυψη των αρμοδιοτήτων των διαφόρων θεσμών ε, ποτέ δεν την κατάλαβα. Υπάρχουν τόσες πολλές προσκλήσεις, τόσα πολλά προβλήματα ανθρωπινών δικαιωμάτων που υπάρχει δουλειά για όλους. Δεν βλέπω ποιος είναι ο... Γιατί να πρέπει το Συμβούλιο της Ευρώπης να κάθεται στη γωνιά του και εμείς στην, ε, από τη Βιέννη στην άλλη γωνιά και να κάνει ο καθένας το δικό του. Αντιθέτως, θα έπρεπε να βρούμε ε, με ποιον τρόπο μπορούμε να βελτιώσουμε τη συνεργασία και να αλληλοσυμπληρωνόμαστε. Το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει την δυνατότητα να εμβαθύνει σε πολλά θέματα και συνεργαζόμενοι μαζί του θα μπορούσαμε να ε, προωθήσουμε μεταρρυθμίσεις. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, πέρυσι το Συμβούλιο της Ευρώπης ε, υιοθέτησε την ε, σύμβαση για την βία κατά των γυναικών, μια πολύ σημαντική σύμβαση η οποία τώρα έχει ανοίξει προς από τα κράτη-μέλη του. Αυτή τη στιγμή η Φορέας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ολοκληρώνει την έρευνα ε, που διεξήγε σε πάνω από 40.000 γυναίκες σε όλα τα κράτη-μέλη ε, θύματα βίας κατά των γυναικών, ε, είτε κατά την παιδική τους ηλικία, είτε θύματα παρακολούθησης. Μια τεράστια συλλογή δεδομένων, η μεγαλύτερη ποτέ στην Ευρώπη, ολοκληρώνεται λοιπόν τώρα και είναι η πρώτη συγκριτική έρευνα ε, στην Ευρώπη που έγινε ποτέ. Είχαν γίνει παρόμοιες έρευνες σε εθνικό επίπεδο, αλλά όχι ποτέ σε, ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτή η έρευνα θα μπορέσει να βοηθήσει το Συμβούλιο της Ευρώπης να πιέσει τα ε, μέλη του να επικυρώσουν την ε, σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και επίσης θα βοηθήσει και τα ίδια τα κρατημέλη όταν θα αφού επικυρώσουν τη Σύμβαση τη Κωνσταντινούπολη, προσπαθήσουν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, θα έχουν πρόσβαση σε συγκριτικά δεδομένα από τι υπόλοιπε χώρε. Ένα ακόμα παράδειγμα είναι η συνεργασία μεταξύ των φορέων. Για παράδειγμα, συνεργαζόμαστε με το Κέντρο Ελέγχου λιμόξεων στη Στοκχόλμη. Ε, θα με ρωτήσετε είναι, ποια είναι η σχέση θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελέγχου λοιμόξεων. Ε, έχουν διαπιστώσει, διαφάζοντας από τις εκθέσεις του Φορέα Ανθρωπινών Δικαιωμάτων, ότι πολύ συχνά είναι η παράτυποι μετανάστες εκείνοι που δεν έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, είτε για λόγους διακρίσεων, είτε για από έλλειψη γνώσης ή οτιδήποτε. Αυτό όμως είναι ένα θέμα ε, ελέγχου λοιμόξεων, ένα θέμα δημόσιας υγείας όταν κάποιες περιφερειοποιημένες ομάδες δεν έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας που χρειάζονται. Και μάλιστα στη συνεργασία με ένα κράτος μέλος ε, κάναμε μια κοινή έρευνα και μια κοινή αποστολή όταν διαπιστώσαμε σε συνεργασία με το φορέα στο Στοκχόλμη ότι υπήρχαν σημαντικά θέματα ανθρωπινών δικαιωμάτων ε, στην έξαρση μιας λοιμόδους νόσου στο κράτος αυτό. Επίσης προσπαθούμε να συνεργαζόμαστε και με άλλους φορείς που ε, διαστηριοποιούνται στον τομέα της ε, εσωτερικών υποθέσεων και της ασφάλειας και της δικαιοσύνη. Προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε πρόσφατα μια ομάδα εργασίας στην οποία συμμετέχει η Europol, η CIPOL και η Frontex. και να συλλέγουμε στοιχεία από αυτούς για την τρέχουσα κατάσταση, αλλά και να βρούμε με ποιον τρόπο μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε στο μέλλον. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα τελευταία 5-10 χρόνια υπάρχει μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Έχει αυξηθεί η συνεργασία και η αλληλεπίδραση μεταξύ αυτών των ε, φορέων που τελικά ε, καθορίζουμε το ευρωπαϊκό τοπίο στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Νομίζω ότι ε, θα ολοκληρώσω εδώ τις παρατηρήσεις μου. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Μπορούμε να φτάσουμε στο τέλος αυτού του τμήματος της τη συνεδριασή μα ξέχασα κάποιον που ήθελε να μιλήσει. Όχι. Τότε από τη δική μου πλευρά απλώ θέλω να κλείσω λέγοντα ευχαριστώ σε όλου σα επειδή ήρθατε με τόσες ενδιαφέρουσες ιδέες για το τι μπορούμε να κάνουμε περαιτέρω, πώς μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά πράγματα και νομίζω και από τη δική μας πλευρά ελπίζω ότι ήταν ενδιαφέρον το ότι η στρατηγική και το σχέδιο δράσης, το νέο πακέτο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η δημιουργία ενός νέου φορέα με τον ειδικό εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό ήταν ένα πολύ σημαντικό θέμα συζήτηση γιατί η πρόθεσή μας ήταν ακριβώς να έρθουμε να έρθει πιο κοντά στην προσοχή σας το γεγονός ότι έχουμε ένα σχέδιο δράσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ελπίζουμε ότι αυτό θα το μεταφέρετε και στο εθνικό επίπεδο με τους ε, συναδέλφους σας και να δείτε πώς μπορείτε να συνδέσετε το δικό σας εθνικό έργο με το πακέτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να κάνετε να ασκήσετε και πίεση στις κυβερνήσεις σας όταν έχονται στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μπορείτε να επηρεάσετε το πώς δρούν στην ΚΟΧΟΜ. Ευχαριστώ λοιπόν. Ευχαριστώ και τις γραμματείες των επιτροπών μας και θα συνεχίσουν αυτές οι επαφές μεταξύ εκπροσώπου για τα ανθρώπινα δικαιώματα πολιτικό σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Όπως ξέρετε όμως το Μάιο έχουμε εκλογές και μάλλον θα έχετε διαφορετικούς συνομιλητές του χρόνου, αλλά όπως και τα προηγούμενα χρόνια θεωρήσαμε ότι αυτή η ανταλλαγή απόψεων ήταν πάρα πολύ καρποφόρα και χρήσιμη. Και τώρα δίνω το λόγο στον συνάδελφό μου, τον κύριο Λόπες Αγγιλάρ. Σας ευχαριστώ κύριε Λοχμίλερ και ευχαριστώ και Διευθυντή του Φορέα για, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την κυρία Βασιούτε για τη δήλωσή της. Ακούσαμε για όλα αυτά τα θέματα που μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα. Ήταν ενδιαφέρουσες όλες οι παρεμβάσεις που ακούσαμε και θα ήθελα απλώς να πω ότι καταρχήν η ρήτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι εδώ για να παραμείνει όταν έχει να κάνει με τη δημιουργία του ενιαίου χώρου φιλε... ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης και το πρόγραμμα της Στοκχόλμης, το πενταετές αυτό πρόγραμμα, το οποίο έχει σε στόχο να αναπτύξει περαιτέρω τις φιλοδοξίες που έχει διακηρύξει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό το σημαντικό τομέα της συνθήκης Λισαβόνας, θα πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί και τούτων λεχθέντων. Είναι γεγονός ότι αυτά τα οποία αναφέρονται σε αυτό το κεφάλαιο της Συνθήκης Λισαβόνας θα πρέπει να πάρουν σάρκα και οστά. Θα πρέπει να προσδιορίζουν όχι μόνο την νομοθεσία η οποία εγκρίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Γι' αυτό έχουμε υποστηρίξει ένα πολιτικό κύκλο συνεργασίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων, δηλαδή μεταξύ ημών με ηττα και ημών με ύψιλον, με τον τρόπο αυτό μπορούμε να εφαρμόσουμε καλύτερα τη στρατηγική μας για τα θεμελιώδη δικαιώματα στο πλαίσιο της νομοθεσίας η οποία αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό σε ό,τι αφορά την χορήγηση ασύλου, την προστασία των εξωτερικών ε, σύνορων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα θέματα λαθρεμπορίας ατόμων, αλλά επίσης και την εκπόνηση νομοθεσίας στο ποινικό δίκαιο και επίσης και την δικαστική συνεργασία. Όλα αυτά σημαίνουν ότι θα πρέπει να οικοδομήσουμε μια νομική κοινότητα με κοινέ αξίες που να περιέχει τη δέσμευσή μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, μια πραγματική κοινότητα αξιών και αυτό θα επηρεάσει και τον τρόπο με τον οποίο, με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τρίτες χώρες. Η ρήτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων όταν διαπραγματευόμαστε συμφωνίες οποιασδήποτε μορφής πολιτικής, διπλωματικής αλλά επίσης και οικονομικού χαρακτήρα και εμπορικού χαρακτήρα με τρίτες χώρες όταν δεν τηρούνται οι προδιαγραφές μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αυτές οι συμφωνίες δεν θα πρέπει να εγκρίνονται. Δεν θα πρέπει να είναι αντικείμενα συμφωνίας. Και όταν οι συμφωνίες αυτές τίθενται σε ισχύ, θα πρέπει πάντα να εποπτεύουμε και να επαγρυπνούμε για την σωστή εφαρμογή της ρήτρας ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έτσι, η ευρωπαϊκή διπλωματία είναι απόλυτα προσιλωμένη στην σε, στην τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλες τις διαδικασίες συνεργασίας. Και όταν ζητάμε θέματα ε, πολύ μεγάλης πολιτικής σημασίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διακυβεύεται και η αξιοπιστία μας σε ό,τι αφορά τη ρήτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων με τα τρίτα, τα τρίτα τους τρίτους, ε, τρίτες χώρες. Εδώ πρέπει εμείς να τονίσουμε την αποφασιστικότητά μας για την προστασία των θεμελιωδών ελευθεριών και των <clears throat> ανθρωπίνων δικαιωμάτων, γιατί, και εδώ καταλήγω, όλα αυτά είναι μια ανοιχτή και διηνεκής διαδικασία, ατέρμον διαδικασία, μη δυνάμενοι εμείς να θεωρήσουμε κάτι δεδομένο, την επίτευξη ενός κράτους δικαίου και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε εκτό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι απλό, δεν είναι ότι μπορούμε να πούμε μα όλοι είμαστε δημοκράτε, έχουμε όλοι τα ανθρώπινα δικαιώματα στα συντάγματά μα οπότε δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα άλλο. Δεν μπορούμε να τα θεωρήσουμε όλα αυτά δεδομένα ότι μπορούμε να θεωρούμε ότι τα δικαιώματα των πολιτών είναι εξασφαλισμένα και όταν συνάπτουμε συμφωνίες ότι δεν υπάρχει τίποτα να συζητήσουμε αν πρόκειται για δημοκρατικές χώρες. Όχι, πάντα υπάρχουν προβλήματα και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι παραμένουμε πιστοί στις αξίες μας, ότι βρισκόμαστε στο ύψος των προτύπων μας και ότι με έναν τρόπο συλλογικό και συνεργατικό μέσα σε ένα ανοιχτό πλαίσιο συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων δια, διαμορφώνουμε μια πολιτική με την οποία θα εξασφαλίσουμε ότι όλα αυτά τα θέματα παραμένουν ενεργά και σημαντικά στην καθημερινή μας ζωή και γι' αυτό εκτιμάμε και το έργο των μη κυβερνητικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, όλων αυτών οι οποίοι ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων αυτών που ακούσαμε σήμερα. Και φυσικά εκτιμούμε ιδιαίτερα το ρόλο του Φορέα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκπροσωπείται από τον κύριο Κιέρομ, τον διευθυντή του. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν παρόντες σε αυτό τον πρώτο γύρο συζητήσεων και περνάμε τώρα στον δεύτερο γύρο θα ξεκινήσει στις 5. Σε 5 λεπτά. Αλλά δεν ξέρω αν έχουν έρθει καλεσμένοι μας ακόμα. Ήρθαν. Α, ωραία. Τότε δεν πρέπει να χρονοτριβούμε και να ζητούμε διάλειμμα λίγων λεπτών. Μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο πάνελ έχοντας ευχαριστήσει το προηγούμενο πάνελ και καλούμε τον κύριο Κασαρίνο το πάνελ που είναι επικεφαλής πλατφόρμας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου στη Φλωρεντία. Είναι ο πρώτος ο οποίος θα λάβει το λόγο εδώ. Και επίσης χαιρετίζουμε την κυρία Μαρίνα Σράμα, Σραμ, λοιπόν, από το Διεθνή Φορέα για την μετανάστευση. Ελάτε παρακαλώ. Και την κυρία Ελέν Σούπιος Νταβίτ για την επαναπροώθηση, τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες. Παρακαλώ. Καλώς ήρθατε.